Έχουμε έξι ψηφίσματα τα οποία έχουν κατατεθεί. Έχει τελειώσει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα αρχίσει τώρα. Ερχόμαστε καταρχήν για τα ψηφίσματα για τον Μπαγκλαντές. Υπάρχει ένα κοινό ψήφισμα. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο, την παράγραφο 8, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Δεκτή. Παράγραφο 9, αρχικό κείμενο. Ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη η I, ε, λατινικό, εδώ υπάρχει μια προφορική τροποποίηση από τον κύριο Τάνοκ, αλλά δεν είναι εδώ ο κύριο Τάνοκ. Θα αναγκαστούμε να ψηφίσουμε χωρί αυτή την ε, πρόταση. Το αρχικό κείμενο λοιπόν ψήφι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας κρίση. Περνάμε στο ψήφισμα για το Κατάρ. Υπάρχει ένα κοινό ψήφισμα τεσσάρων ομάδων. Ψηφίζουμε καταρχήν την παράγραφο 8, το αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Δεν ήταν πολύ σαφές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Απολύτω, συγγνώμη. Αιτιολογική σκέψη Β. Και εδώ ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσανε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Ε ηλεκτρονικά και πάλι άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο, όπως έχει τροποποιηθεί, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέλος, το ψήφισμα στην ε, δίκαια δίκη στην ε, Βολιβία, περίπτωση του Ελότο Ασό και Μάριο υπάρχει ένα κοινό ψήφισμα τεσσάρων ομάδων. Η τροπολογία 4, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο με μια προφορική τροπολογία της κυρίας Δεκαίζερ. Και αυτή θα ψάχνει. Δεν τη βρίσκω. Στο άρθρο 4 να βγουν οι λέξεις να αναλυφθούν συγκεκριμένες ενέργειες και βήματα από την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων λέει, να πάρει συγκεκριμένα βήματα αλλά και πράξεις και ενέργειες. Αντιρρήσεις. Είναι επαρκής οι αντιρρήσεις. Οπότε δεν μπορεί να γίνει δεκτή η προφορική αυτή ε, τροποποίηση. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 4 ψηφίζουμε ψήφι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μετά την αιτιολογική σκέψη α, τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται μετά την ε, G, τροπολογία 2, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, το σύνολο με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρακτικά της συνεδρίας αυτής θα εγκριθούν στην επόμενη συνεδρία του Κοινοβουλίου και τα ψηφίσματα αυτά θα διαβιβαστούν στους ε, αποδέκτες τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εύχομαι σε όλους τους βουλευτές και τους υπαλλήλους μια καλή επιστροφή. Α, ο κύριος Όντι για διαδικαστικό θέμα προηγουμένως.